αλλά Abdel Fattah και μπορούμε να περάσουμε στις πληροφορίες. Καταρχήν θα ψηφίσουμε για, τα 6, για τις έξι προτάσεις ψηφίσματος για το Ιράν. Τροπολίγια παρθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ξεχρήβωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Συμπεριλαμβάνουμε και τον κύριο ταβαρέ που δεν βρίσκει τη, το κουμπί, την κάρτα του. Ωραία. Ε, κλείσε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμφωνείτε. Ωραία. Μπορούμε να ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολο του υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στα έξι προτάσεις ψηφίσματος για την Αίγυπτο. Ιδιαίτερα την περίπτωση του blogger αλλά Αμπτελ Φατά. Ε, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Κύριε Μακοβέη, διαδικαστικό. Η ψήφος μου είναι θετική. Υπερψήφισα το κείμενο. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Ωραία. Εντάξει, καταγράφηκε. Αυτά για τις πληροφορίες. Ε, τα... Τα πρακτικά